δεν θα ήταν σωστό, για παράδειγμα, να απαγορεύσουμε τα ε, χάρτινα κυπελάκια επειδή περιλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό πλαστικών. Και πρέπει να βρούμε πάντα εναλλακτικέ λύσει, βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έρκα Αντρίου. Ένα λεπτό. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία για την εξαίρετη αυτή έκθεση. Ε, το θέμα επίγει. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε κίνδυνο έχουμε δημιουργήσει μια έβδομη ήπειρο με 80.000 80 ε, εκατομμύρια τόνους πλαστικών. Θα πρέπει να ξαναδούμε το οικονομικό μας μοντέλο. Γιατί κινδυνεύει το μέλλον των, βιοσυστημάτων μας. Ε, θα πρέπει να μειώσουμε δραστικά την χρήση του πλαστικού στην Ευρώπη και να εφαρμόσουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει ταχύτητα να βγούμε από την νεοφιλελεύθερη λογική που μας οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη κατανάλωση και μολύνει τον πλανήτη. Τέλος, θα πρέπει να είμαστε λογικά συνεπείς με τον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε ένα κείμενο το οποίο επιστεί την προσοχή στην μόλις από τα πλαστικά. Και αυτή τη στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε πλαστικά μπουκάλια και πλαστικά καλαμάκια. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, να σταματήσουμε τη χρήση αυτών των αντικειμένων μέσα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σουίτσα. Κύριε Σουίτσα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ζούμε ε, αδιαφεσβήτητα στην εποχή των πλαστικών. Ο το αρνείται. 8 δισεκατομμύρια τόνους πλαστικού έχουμε ε, παράξει σε 65 χρόνια. Πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Καλωσορίζω το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου και ελπίζω ε, αύριο αυτό να ολοκληρωθεί και με μια ικανοποιητική ψηφοφορία. τα περισσότερα πλαστικά που χρησιμοποιούμε είναι μιας χρήσης, τα μισά και πλέον. Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις και όπου υπάρχουν αυτές θα πρέπει να ε, τις χρησιμοποιούμε ως υποκατάστατα των πλαστικών. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μέσω έρευνας και καινοτομία για να βγουν και νέα προϊόντα στην αγορά. Υποστηρίζω απολύτως αυτή την πρωτοβουλία και την οδηγία και ελπίζω να εφαρμοστεί το συντομότερο και να μεταφερθεί στην νομοθετία μας. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ ο κύριος Χάνσεν. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς το μικρόφωνο το μιλητή σταματάει. Yes, please turn your microphone. Is it on now? Thank you. Κάποιο πρόβλημα έχει το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Ε, κοινωνία καταναλωτική. Έχουμε, παίρνουμε ένα καφέ για το δρόμο και το πετάμε μετά το κυπελάτι. Καμιά φορά χρειάζονται απαγορεύσεις για να κοπούν οι κακές συνήθειες. Ε, υπάρχουν ε, υποκατάστατα. Εγώ θα ήθελα μεγαλύτερη φιλοδοξία όμως για την ευθύνη των κρατών μελών και πολύ πιο δραστική μείωση και με τις συσκευασίε. Δυστυχώς αυτό δεν πέρασε. Χάσαμε την ευκαιρία αυτή. Πριν από ένα μήνα για πρώτη φορά έγινα πατέρας και θέλω να κοιτάζω κατάματα το γιο μου και να μπορώ να του λέω με καλή τη συνείδηση ότι κάναμε κάτι για να διατηρήσουμε το πλανήτη μας βιώσιμο και για τα παιδιά μας. Είναι ένα μόνο βήμα, το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το αγοράκι σας, το νεογέννητο. Ε, διαδικασία ΚΑΣΔΙΑΕ. Εάν ε, τηρήσετε το μονόλεπτο, θα πάρετε το λόγο όλοι όσοι το ζητήσατε. Κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε η πρώτη γενιά πολιτικών που καταλάβαμε τι ζημιά κάνουμε στο περιβάλλον με τα πλαστικά μιας χρήσης και είμαστε και η τελευταία γενιά όσων μπορούν κάτι να κάνουν γι' αυτό. 75% αυτού του είδους προϊόντων καταλήγουν στις θάλασσές μας. Εγώ είμαι από τη Μάλτα και από τον Κόντζο. Και τα ξέρω αυτά γιατί έχουμε δει τεράστιες εκτάσεις πλαστικών κοντά στις ακτές μας και αυτά βέβαια καταλήγουν και στα στομάχια των ε, ψαριών που καταναλώνουμε. Ε, θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα πλαστικά. Και ακόμη και που μέχρι το 2021 θα χρειαστεί να περιμένουμε για να παγορευτούν. κάτι είναι κι αυτό. Ε, θα πρέπει όμως να αρχίσει ο καθένας από την ατομική του ευθύνη. Ε, αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς για να αλλάξει τις συνήθειές του, κάνει διαφορά. Δεν έχουμε πλέον χρόνο και πρέπει να αναλάβουμε δράση αμέσω. Ευχαριστούμε κυρία Γόρντ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συνολική ποσότητα απορριμμάτων αυξάνεται διαρκώ σε παγκόσμια κλίμακα. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 3,5 τόνοι κατά κεφαλή ε, παράγονται ετησίω. Πάνω από 400 ε, κιλά ε, Ετησίω ανά άτομο σε οικιακά ε, απόλυτα. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2030. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει πραγματική αποσύνδεση μεταξύ, της, ε, μεταξύ των αποβλήτων και της διαχειριστή τους και της οικονομίας μέχρι το 2020. Τα πλαστικά είναι το 1 τέταρτο όλων των απορριμμάτων που βρίσκονται στις θάλασσες και στις ευρωπαϊκές ακτές. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ερχόμαστε από 28 διαφορετικές χώρες, αλλά έχουμε ένα είδη ίδιο κοινό μάλλον σπίτι, μια κοινή αστεία. Τον πλανήτη Γη. Οι νέοι το γνωρίζουν αυτό και μπούχτησαν. Μπούχτησαν και απαιτούν να αλλάξουμε εμεί. Ζητώ λοιπόν από όλου σα να υποστηρίξετε τι κλιματικέ του απεργίε, τι παρασκευέ του μέλλοντος όπω τι έχουν ονομάσει. Γιατί εάν δεν σταθούμε στο πλευρό του, δεν θα μα εκλέγουν και εκείνοι στο μέλλον. Ευχαριστούμε ο κύριος Φλάναγκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλάμε για έναν τομέα εδώ όπου θα πρέπει να αναλάβει πραγματικά δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μόνες τους. Ακούω συχνά αυτή τη φράση πέτατο είναι μια φράση την οποία πρέπει να την παύσουμε, να την αλλάξουμε. Όταν λέμε σε πολλές περιπτώσεις πέτατο, εννοούμε ότι πήγε στο καλάθι των αχρήστων, ότι έφτασε, πήγε μετά στη σκουπιδιάρα και κάπου κατέληξε. Η πραγματικότητα είναι πουθενά δεν κατέληξε. Διότι αυτό ε, που συμβαίνει είναι ότι το κάθε πραγματάκι που χρησιμοποιούμε πρέπει να διερωτόμαστε όταν το πετάμε. Πού κατάληγει. Δεν μπορούμε απλώς να μένουμε όμως σε αυτή την ερώτηση. Οι εταιρείε που παράγουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει επίσης να θέτουν την ερώτηση στον εαυτό τους και θα πρέπει να αναγκαστούν να ρωτούν τους εαυτούς τους. Πραγματικά ε, είμαι περήφανος για τους νέους και τη δουλειά που κάνουν. Θα πρέπει όμως και τις γιαγιάδες μας και τις προγιαγιάδες μας να τις επενέσουμε γιατί γνώριζαν την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος πριν επινοηθούν αυτοί οι όροι. Διότι ε, ζούσαν αναγκασμένες να τα πράττουν αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάλφοι, και εγώ στηρίζω αυτή την συμφωνία που επιτεύχθη στον τριμερή διάλογο και χαίρομαι που την υποστηρίζουν και, και την υποστηρίζει μια ευρία γκάμα πολιτικών ομάδων. Θα μας βοηθήσει να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να εξοικονομήσουμε και φυσικού πόρου, διότι δεν είναι ανεξάντλητοι. Θα πρέπει πάντοτε να επιλέγουμε προϊόντα τα οποία δεν ε, ε, είναι συσκευασμένα σε πλαστικό. θα πρέπει όλοι και ο καθένας από εμά να συνεισφέρουμε. Και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε σε τέτοιου είδους κλίμακα πλαστικά μπουκάλια. Αυτή η οδηγία άλλωστε καθιστά, ε, δημιουργεί υποχρεώσεις και για τους παραγωγούς. Η τσεχική δημοκρατία είναι μια χώρα στην οποία ε, ανακυκλώνουμε πάρα πολύ. 42% των αποβλήτων μας ε, των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής ανακυκλώνονται σε εμάς 62%. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Okay. Φαρία, ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την πρόταση αυτή της οδηγίας έχουμε ήδη αναλάβει ευθύνες. Η στατικική για τα πλαστικά για τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε ε, θα πρέπει σε όλα τα τελικά προϊόντα να προσέχουμε τι γίνεται με τη σύσταση και να μην καταλήγουν όλα αυτά στους ωκεανούς και καταστρέφουν το περιβάλλον και τη βιοσφαίρα. Όλα τα απορρίμματα που βρίσκονται στους ωκεανούς έχουν πρόλευσή τους εδώ στην ξηρά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπευθυνότερη κατανάλωση, ευφιέστερη, και να αναλάβουμε τα κατάλληλα οικολογικά μέτρα και ευθύνε. Η πρόταση τη Επιτροπή ΕΝΒΗ, ε, οι πλαστικέ σακούλε που είναι πολύ ελαφρύ να ε, περιληφθούν στον κατάλογο απαγόρευση δεν πέρασε. Όμω θα πρέπει εδώ πραγματικά να γίνει μια σωστή αποσύνδεση τη ε, διαλογή και του τι καταλήγει στους ωκεανούς είτε είναι υλικά βιοδιασπόμενα, είτε είναι υλικά που μπορούν να καταλήξουν σε κάψη, πρέπει να μην επιτρέπονται. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα που προβλέπει η οδηγία με φιλόδοξου στόχου που να του επιδιώξουν ε, χωρί ε, πάυση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δρογεύς. Ευχαριστώ. Ε, πρέπει να σας πω από την αρχή ότι δεν είμαι οικοτρομοκράτης, αλλά δεν ξέρω αν είμαι και πάρα πολύ ε, υπέρ αυτής της πρόταξης, της πρότασης. Πρέπει να σας πω ε, ότι δεν ε, με ικανοποιεί πάρα πολύ η συζήτηση. Υπάρχει κάτι που χάνουμε. Υπάρχουν ε, πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε ένα οδικό χάρτη και ένα πρόγραμμα ε, με μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Τι πρέπει να κάνουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Με τη σειρά. Βεβαίως, οι καταστάσεις είναι περίπλοκες, αλλά δεν έχουμε ένα σύνολο που πρέπει να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα. Χρειάζεται συνέχεια δικαίου στα διάφορα κράτη και συγκεκριμένες διαδικασίες για να καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα. Καλή είναι η ευαισθητοποίηση, αλλά δυστυχώς εμείς δεν είμαστε συνεπείς ε, στην επιβολή κυρώσεων και προστήμων για εκείνους που ρηπαίνουν τον πλανήτη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και τελευταίο στη διαδικασία Κάρσια, κύριος Σον Κέλλη. Παρακαλώ. Ε, συζητήθηκα το θέμα αυτό και στην Επιτροπή Αλίας εδώ και αρκετό καιρό και χαίρομαι για την έκβασή του. Η Επιτροπή, στην Επιτροπή Αλίας εξετάσαμε το θέμα εξαιτία του γεγονός ότι πολλά από τα πλαστικά βρίσκονται στη θάλασσα και μάλιστα καταλήγουν στις κοιλιές των ψαριών. Επίσης έχουμε το φαινόμενο των ε, χαμένων απολεσθέντων ε, εργαλείων, αλλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα. Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε γρήγορα. Ε, πολλά από τα πλαστικά μονή χρήση μπορούν να αντικατασταθούν, για παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ απλό. Όμω, μακροπρόθεσμα, στέλνουμε και ένα μήνυμα στη βιομηχανία ότι η μόλυνση από τα πλαστικά θα πρέπει να σταματήσει και τα πλαστικά θα πρέπει να συλλέγονται και να επαναχρησιμοποιούνται ή να κυκλώνονται. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να δώσουμε τέρμα στη μόλις του περιβάλλοντο από τα πλαστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Τίμερμανς, μόνο της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούγοντα τι ομιλίε των Ευρωβουλευτών, σκεφτόμουν πόσο μοναδικό είναι το ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν με αυτή την πρόταση με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα από την δεξιά μέχρι την αριστερά. Γιατί φτάσαμε τόσο γρήγορα εδώ. Γιατί νομίζω ότι ήταν γρήγορη διαδικασία. Αν γυρίσουμε πίσω 3-4 χρόνια δεν μας φαινόταν θα λήξει τόσο γρήγορα το θέμα. Ε, και Εκτός του να συγχαρούμε τους, την συγκέντρα και του ε, σκιώδες θα πρέπει να συγχαρούμε και όλους του υπόλοιπου οι οποίοι ενέπνευσαν και την κοινωνία και τι ευαισθητοποίησαν έναντι του ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ επίγον και κρίσιμο. Η Έλλη Μακάρθρο, ας πούμε, που ήταν από τους πρώτους που... Ε, ε, ευαισθητοποίησαν το κοινό. Ε, είχαμε ψηρές και ντοκιμοντέρ στην τηλεόραση, στα μέσα ενημέρωσης, ε, το, τα ντοκιμοντέρ του Άτεμπορο για παράδειγμα. Η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δημιούργησαν όλο αυτό το κλίμα, ο καθημαϊκό κόσμος, το κλίμα αυτό στην κοινωνία του, του, του, του επίγοντος. Θα πρέπει λοιπόν να συγχαρούμε και όλους αυτούς που είναι εκτός της πολιτικής και που μας βοήθησαν. Θα συμφωνήσω όμως με, με, με αυτούς από εσά που είπαν ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Ας μην είμαστε απλώς αυτάρεσκοι. Να θυμόμαστε ότι ο δρόμος είναι μακρύς μπροστά μας, μέχρι ότου εξασφαλίσουμε την κυκλική οικονομία. Αυτό όμως είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι ένα μοναδικό βήμα επίσης επειδή ε, κλείνει το κύκλο του πλαστικού και αναγνωρίζεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ασιατικές χώρες ενδιαφέρονται πολύ για αυτό που κάνουμε. Οι λατινοαμερικανικές χώρες επίσης. Οπότε, παρόλο ότι το δικό μας μερίδιο της μόλυνση είναι σχετικά περιορισμένο, η αλλαγή του οικονομικού μας μοντέλου έχει παγκόσμιες επιπτώσεις και θα αλλάξει τα οικονομικά μοντέλα και αλλού. Οπότε μην αποθαρρύνεστε από τις φωνές που λένε ότι η Ευρώπη αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό το μέγεθος της οικονομίας μας είναι τέτοιο που αν αλλάξουμε το δικό μας οικονομικό μοντέλο, το κάνουμε πιο βιώσιμο, θα αλλάξουμε και το οικονομικό μοντέλο αλλού στον κόσμο. Και συμβαίνει αυτό ήδη. Η μόλυνση από τα πλαστικά ε, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές χώρες και περιοχές του κόσμου. Και θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξή. Όλα αυτά θα επηρεάσουν και τις συσκευασίε. Γιατί περιλαμβάνονται οι, οι, οι, ε, στην πρότασή μα Μέχρι το 2030 θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμε. ανακυκλώσιμες. Επίσης, τα μικροπλαστικά είναι τρομακτική απειλή για την υγεία μα. Θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα προϊόντα στα οποία δεν χρειάζονται, για παράδειγμα τα απορριπαντικά ή τα καλλιντικά, αλλά μετά θα πρέπει να δούμε και τα προϊόντα στα οποία χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, τα μικροπλαστικά, για παράδειγμα τα λάστιχα αυτοκινήτων, που είναι πολύ μολυσματικοί παράγοντες. Μην ανησυχείτε, θα, το, θα γίνει αυτό στην επόμενη Κομισιόν, όποια και είναι η σύστασή της. Είναι κάτι στο οποίο επιμένουν όλοι εδώ. Και γι' αυτό το λόγο θα αποτελέσει και μέρημνα Τη επόμενη Κομισιόν, του επόμενου Συμβουλίου και του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την προσήλωσή σας και τη δεσμευσή σας, κύριε Τίμερμαντ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρή, στην εισηγητριά μα. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Δύο λόγια μόνο θα πω. Πραγματικά, μαζί. Αυτή είναι η λέξη κλειδί μαζί θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το σύνολο ε, των συναδέλφων που μας υποστήριξαν με δύο ε, ε, εξαιρέσεις του συναδέλφους του Brexit που καλά θα κάνανε εδώ να λυπούνται και να θλίβονται για τις θέσεις εργασίας που χάνονται στη Βρετανία από το Brexit. Εν πάση περιπτώσει. Τι είχε πει ο Τζον Φιτζέραλτ Κέννεντι το 1963 στην Ουάσιγκτον ότι τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο και μπορούμε να τα λύσουμε. Οι δυνατότητές μας δεν γνωρίζουν όρια. Χωρίς ε, όρια λοιπόν κανένα ανθρωπογενές πρόβλημα δεν μπορεί ε, ε, παρά να ξεπεραστεί από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κινητήρια δύναμη για τη λύση είναι μια, μια πρώτη αυτή ε, προσπάθεια, αλλά είμαστε όλοι καθοδόν και εμπρός, για να αναφερθώ και σε κάτι που καταλαβαίνετε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει εδώ αυτή η συζήτηση και στις 5 ώρα θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Προχωρούμε, συνάδελφοι, στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη, το οποίο είναι η ε, έκθεση του κυρίου Τσουρκάνου, ε, για ε, τα λοιπάσματα ε, που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, για τέσσερα λεπτά το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Τσουρκάνου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδεις εισηγητές και αγαπητοί συντάκτες γνωμοδότησης, νομίζω ότι κάναμε καταπληκτική δουλειά. Καταφέραμε από κοινού να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή στη διάρκεια της παρούς κοινοβουλευτική περίοδου. Είναι το αποτέλεσμα της δικής σας δουλειάς, της δικής μου δουλειάς, ε, γεωργών, ε, εργαζομένων στον κλάδο, παραγωγών, λοιπασμάτων. Συμμετείχαμε όλοι και συνεισφέραμε όλοι στην προσπάθεια αυτή είναι ε, σωστή η έκθεση, συνεπής και βοηθάει όλα τα μέρη. Δύο χρόνια χρειάστηκε να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας, τους αγρότες μας και σήμερα δρέπουμε τους καρπούς. Βλέπουμε τα αποτελέσματα και περιμένουμε την ψήφο εμπιστοσύνη σα. Ήταν εντατικέ οι διαπραγματεύσει με τρει προεδρίε, παρακαλώ, εσθονική, βουλγαρική, που φτάσαμε στο παραπέντε ε, για να καταλήξουμε. Και ολοκληρώσαμε τον τέταρτο τριμερή διάλογο επί Αυστριακή Προεδρία πέρσι τον Νοέμβριο, όπου δείξαμε ότι μπορούμε και συμβιβασμού να κάνουμε όταν πρόκειται για συνένεση. Θα ήθελα επ' ευκαιρία να ευχαριστήσω πραγματικά την Αυστριακή Προεδρία. Ήταν πολλέ οι εντάσει και οι τριβέ αλλά και οι συγκινήσεις στις διαπραγματεύσεις. Ε, και όποιος νομίζει ότι ήταν εύκολο το θέμα, πλανάτε Πλάνιν ή τραν. Πρέπει να σας πω ότι μετά την έκθεση αυτή ε, και αφού τεθεί σε ισχύ νομοθεσία, όλοι οι ενεχόμενοι και στη Γεωργία αλλά και οι καταναλωτέ θα υποφεληθούν. Διότι ο νέο κανονισμό που έρχεται να αντικαταστήσει τον παλαιό πρόκειται να ανοίξει την εσωτερική αγορά για κάθε είδου λοιπάσματα είναι τμήμα του πακέτου της ε, κεκλικής οικονομίας και αφορά λοιπόν όλα τα είδη των λοιπασμάτων. Εναρμονίζει τα όρια για τους ρηπαντές τα μισά λιπάσματα στην ευρωπαϊκή αγορά σήμερα δεν καλύπτονται από την κείμενη νομοθεσία. Μόλις το 5% των οργανικών λιπασμάτων ή των οργανικών μάλλον προϊόντων ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα. Ε, τι στόχο έχει αυτός ο κανονισμός, το 5% να γίνει 30%. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει πάνω από 6 δισεκατομμύρια τόνους ε, φωσφορικά λιπάσματα ε, ε, και θα μπορούμε να ε, ανακτούμε ε, από την τέφρα ε, της ανακύκλωσης των υπολοιμάτων σφαγίου για να τα χρησιμοποιούμε ως λιπάσματα και να μειώνουμε τον κίνδυνο για τους καταναλωτές και την υγεία τους και το περιβάλλον. Το κάδμιο, ας πούμε, και τα φωσφορικά λιπάσματα Έχουμε 60 μιλιγκράμμ το, το κιλό, ρυθμίζεται, ε, αυτή τη στιγμή στεθεί σε ισχύ νομοθεσία, δηλαδή τρία χρόνια μετά την έγκρισή της. Ε, σύνοψίζω λοιπόν, ε, ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα έχει πιο υγιεινά τρόφιμα, οι Ευρωπαίοι αγρότες θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερα λιπάσματα, ασφαλέστερα, αλλά και σε οργανικά λιπάσματα που θα κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, έτσι ώστε ε, μετά την ανακύκλωση και τη χρήση ε, να ε, προχωρούμε καλύτερα. Και η βιομηχανία θα ε, έχει περισσότερο τη δυνατότητα παροχής πρώτης ύλη. Δεν θα έχουμε μονοπόλια ε, δεν θα έχουμε τεχνητά ακριβέ τιμέ και έτσι θα σωθούν και πολλές θέσει εργασία, εκατομμύρια θέσει εργασία. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Τα κράτη-μέλη ακόμα θα μπορούν να επιβάλλουν εθνικέ προδιαγραφές και πρότυμα για την κυκλοφορία στην αγορά λοιπασμάτων. Επίσης, ε, διατηρείται η δυνατότητα της αμοιβαία αναγνώρισης λοιπασμάτων. Θα πρέπει να κινητροδοτηθούν οι ενδιαφερόμενοι έτσι ώστε να προάγουν καινοτόμα λοιπάσματα χωρίς κάδμιο που θα αποφέρει και οικονομικά αποτελέσματα. Γενικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με την τελική εκδοχή αυτή του κανονισμού. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία μας. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Γκαρντίνη εκ μέρους της Επιτροπής ΕΝΒΗ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι εδώ εργαστήκαμε ε, όσο το δυνατόν συντομότερο και καταλεφ, καταφέραμε να αποσπάσουμε αυτά που θέλαμε. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα παράδειγμα του πώς η υπομονή μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα και μια καλή διαδικασία. Έχουμε ξεκινήσει κάτι σημαντικότατο. Ανοίξαμε την ε, ενία αγορά σε μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που τώρα αποκλείονταν από από τα οργανικά, τα ε, άλλα λοιπάσματα όπως και αν ονομάζονται και το κάναμε μεγάλη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος. Καταφέραμε να θέσουμε μέγιστα όρια, ιδίω για το κάτι που ήταν δύσκολο και ε, πριν δεν υπήρχαν και θέλω να το ε, τονίσω, πριν δεν υπήρχαν και πραγματικά είχαμε το χαμηλότερο όριο παγκοσμίω το χαμηλότερο είναι το διπλό 60 ε, μιλιγκράμμ και φτάσαμε στα 120. Το, χαμηλότερο ήταν αλλού. Ε, ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους για την αφοσίωσή τους ε, και νομίζω ότι κάναμε μια εξαιρετική δουλειά. Ως Ιταλίδα επιτρέψτε, με, επιτρέψτε μου να μιλήσω κυρίως για τις ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις της Ιταλίας που είναι όμως άριστες. Είναι άριστες και θέλουν να εκμεταλλευτούν από το σύστημα της κυκλικής οικονομίας που το είχαν επινοήσει πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καν το αναφέρει. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκαρδίνη. Επόμενο ομιλητή ε, ε, από πλευρά τη Επιτροπή Γεωργία, ο κύριο Χέιτεμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, ε, συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις και σκληρά εργάστηκα για τον νέο αυτό Τώρα επιτέλους μπορούν οι αγρότες και οι κυπουροί να χρησιμοποιούν περισσότερα οργανικά λιπάσματα. Κοπριά, ας πούμε, αντί τα τεχνητά λιπάσματα. Μέχρι σήμερα οι αγρότες δεν μπορούσαν να ε, να χρησιμοποιήσουν ε, όλη την κοπριά που ε, παρήγαγαν ε, για ε, ίδια χρήση είχαν ένα περιορισμό και ό,τι περίσσευε έπρεπε να πληρώσουν για να διατεθεί. Και επίσης δεν μπορού, έπρεπε να εισάγουν ανόργανα λοιπάσματα. Είναι πραγματικά τρομερά αυτά τα πράγματα στη χώρα μου. Χρησιμοποιούμε πολύ φυσικό αέριο και τα οργανικά λιπάσματα είναι προϋπόθεση για το υγιεινό έδαφος έτσι ώστε να παράγει περισσότερο η γεωργία και να έχουμε ε, καλά φυτά ε, ε, και επίσης ε, διατηρείται και η ποιότητα του εδάφους. Είναι πλούσιο το εδάφος και δεν εκπλήνεται. Ε, είναι αμοιβαία η ωφέλεια λοιπόν. Ήταν ένα πάγιο αίτημα ε, ετών των αγροτών και επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι έχει την ίδια γνώση και σοφία ως οι αγρότες. Ο Αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ο κύριος Τίμπερμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τον κύριο Χάρτσμαν να λέει ότι εργάστηκε σκληρά, η κυρία Γκαρδίνη πολύ, με πολύ συνέπεια. Το αποτέλεσμα φαίνεται. Είναι πολύ καλό. Βελτιώνει το κανονισμό για τα λοιπάσματα. Ευχαριστώ τους ε, εισηγητές του Κάνου, Γκαρδίνη, Χάρτεμα και τους Σκιώδης για όλη την πολύτιμη συνεισφορά σας. Ο κανονισμός συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων κυκλικής οικονομίας, εις ό,τι αφορά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Τώρα καλύπτονται μόνο οι... τα λοιπάσματα απορριχτά. Τώρα θα έχουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα απλουστεύει το νομοθετικό πλαίσιο για τους οργανικού, τα οργανικά λοιπάσματα. Έτσι θα μπορέσει να ανοίξει η ενιαία αγορά σε καινοτόμα προϊόντα από υποπροϊόντα ε, απόβλητα, επαναχρησιμοποιούμενα. Προφανώς θα φροντίσουμε για την ασφάλεια ε, της υγείας και του περιβάλλοντος. Ε, αυτό θα ωφελήσει πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. τα οργανικά λιπάσματα είναι το 50% της αγοράς και έχουν μεγάλο δυναμικό, μπορεί να γίνει βιώσιμη, αποδοτική η γεωργία οι αναδυόμενε επιχειρήσεις να ωφεληθούν. Με την ψήφο σα σήμερα τα προϊόντα αυτά θα ενταχθούν στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και θα υπάρχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Παράλληλα αυτός ο κανονισμός δίνει και διασφαλίσει για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επίσης θα βάλει και όρια υποχρεωτικά για το ενικό το κάδμιο κυρίως ε, τον υδράργυρο. Τώρα έχουμε κοινά όρια για το κάδμιο. Μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής θα δούμε αν τα όρια μπορούν να μειωθούν. Έτσι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, η συμβαστική λύση καλύπτει όλα τα συμφέροντα. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουν όλοι και ο κλάδος λοιπασμάτων της Ένωσης που θα έχει καλύτερη πρόσβαση καινοτόμων προϊόντων στην ενία αγορά και θα είναι και ε, ανταγωνιστικά ως προς το κόστος ε, τα υλικά, οι πρώτες ύλες και βέβαια οι ε, κατασκευαστές και οι γεωργοί θα μπορούν να προστατεύουν τα εδάφη από τοξικά προϊόντα και οι πολίτες θα ωφεληθούν γιατί οι τοξικές ουσίες μειώνουν την ασφάλεια του εδάφους, υπεδάφους, υπογείων υδάτων, τροφίμων. Ε, τα χημικά λιπάσματα μπορεί να αντικατασταθούν και με επεξεργασμένη κοπριά. Αυτό εντάσσεται στο σχέδιο δράση γιατί συμβάλλει στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των θρεπτικών ουσιών για τη γεωργική παραγωγή. Παράλληλα, ε, η Κομισιόν εργάζεται για πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών που δεν πρέπει να μολύνονται και να ε, βλάψουν την υγεία. Η κοπριά δίνει τη δυνατότητα καλύτερης χρήσης των θρεπτικών ουσιών και από άποψη γεωργίας και από άποψη περιβάλλοντος. Γι' αυτό το Κοινό Κέντρο Ερευνών το 2017 ε, ε, έκανε μια μελέτη πειραματική για να δει πώς ε, μπορούμε να αντικαταστήσουμε χημικά λιπάσματα στη γεωργία από κοπριά. Ε, που δεν συνεπάγεται περιβαλλοντικούς κινδύνους ε, που είναι το, ένα βασικό θέμα. Το έργο συνεχίζεται, ένα σχέδιο μελέτης θα παρουσιαστεί κανονικά στο τέλος του 2019. Τα κριτήρια αφορούν τη χρήση των λοιπασμάτων, όχι τη διάθεσή του στην αγορά. Δεν επηρεάζονται λοιπόν από τον κανονισμό για τα λοιπάσματα και δεν θα επηρεάσουν την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Όμως, οπωσδήποτε, είναι ε, πρόσθετη δράση συμπληρωματική για ε, κυκλική οικονομία αποτελεσματική και ασφαλή. Στηρίζομαι απόλυτα τη συμβαστική λύση που ε, ανεβρέθη. Ε, υπολογίζομαι σε εσά ε, για να συμβάλλουμε στο, στη βελτίωση του κλάδου προς το συμφέρον της κυκλικής οικονομίας, της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι ένα συγκεκριμένο ε, βήμα για τους βιώσιμους στόχους και το βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης που γίνεται πιο κατεπήγον σήμερα από ποτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν... Δεν βλέπω τον κύριο Βαγουέσα στην αίθουσα, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπόγκοβιτς, εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, μετά από έναν ε, τριμερή διάλογο και επιτυχής διαπραγματεύσεις ολοκληρώσαμε το έργο μας. κάναμε πολλές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τα ανόργανα λοιπάσματα και τώρα έχουμε νέες προτάσεις για τα οργανικά. Και αυτό συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Ο στόχος είναι ε, τις θρεπτικές ουσίες ε, από τα οργανικά ε, από τις οργανικές ουσίες να μην τις σπαταλάμε. Το, από το προϊόν της κομποστοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλύτερα ως λίπασμα. Μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό σε μεγάλη κλίμακα. τώρα θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις ώστε τα λοιπάσματα αυτά που δρούν, ε, να μην δρούν επιζήμια για το περιβάλλον. Επίσης έχουμε και μια συμβιβαστική λύση για το κάδμιο που είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Υποστηρίζω και το τμήμα εκείνο που ασχολείται με τις καινοτομίες και τις δυνατότητες που δίνονται ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μέχρι τώρα ήταν ε, περιορισμένες ως προς την πρόσβαση στην αγορά. Αυτός ε, ο τομέας αριθμίζεται επίσης. Προφανώς έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά και κάναμε πολλά για την κυκλική οικονομία. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο κύριος Ταραμπέλα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σίγουρα τα λοιπάσματα είναι σημαντικά για τη γεωργία. Η χρήση του όμω μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον και την επιστηστική ασφάλεια. Ιδιαίτερα δεν υπάρχουν ρηπογόνε ουσίε σε αυτά τα προϊόντα λίπανση. Η σωστή χρήση λοιπόν και η ακίνδυνη χρήση των ειδών λίπανση έχει κέρια σημασία για μια βιώσιμη γεωργία, για την προστασία του περιβάλλοντο και για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Και ο κανονισμό για, τα, για τα προϊόντα λίπανση εντάσσεται στο πακέτο τη κυκλική οικονομία, γιατί το σχετικό νομοθέτημα βάζει, ε, ε, δίνει την ίδια μεταχείριση στα κλασικά ανόργανα λιπάσματα μαζί με τα οργανικά λιπάσματα που χρησιμοποιούν ε, πρώτες ύλες ε, που προς το παρόν ε, διατίθενται ως απόβλητα. Σημαντικό μέλημά μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την εγγύηση που δίνουμε στους γεωργούς να αγοράζουν παντού στην Ευρώπη ποιοτικά προϊόντα. Με τους νέους κανόνες διασφαλίζουμε αυτή την ισορροπία και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ώστε να βοηθήσουμε τους γεωργούς να έχουν καλύτερη απόδοση. Πρόκειται για μια κρίσιμη φάση στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα για το κάδμιο. Παρόλο που κάναμε κάποιες προσπάθειες, τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξα από την αρχική θέση της διαπραγμάτευσης που είχαμε υπερψηφίσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξαιτία μια ανασχετική μειοψηφία στο Συμβούλιο δεν καταφέραμε να διαφυλάξουμε τα όρια καδμίου 40 και 20 ε, χιλιοστόγραμμα το κιλό που είχαμε εγκρίνει εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, βέβαια, παρόλα αυτά έχουμε μια πρόοδο για το κάδμιο. Ε, προαιρετική ετικετοθεσία μικρής περιεκτικότητας, ρήτρα επανεξέτασης μετά από τετραετή εφαρμογή, ε, εθνικές εξαιρέσεις για τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν ήδη χαμηλότερες οριακές τιμές καδμίου και μέτρα για την απορρίπαση. Και ευχαριστώ τον συναδελφό Τουρκάνο παρά τις ε, δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις που είχαμε και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους και οδησηγητές Γκαρτίνη, Τωμά και Βαγουένσα για την αγαστή συνεργασία που επικράτησε στις συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα. Ο κύριος Χότ έχει το λόγο, εκ μέρους του ECR. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά είχαμε δραστικές οριακές τιμές ε, ε, περιεκτικότητας φωσφορούχων λιπασμάτων σε κάδμιο. Και αυτό χτύπησε ιδιαίτερα την πολωνική χημική βιομηχανία που είχε την κρούπα αζώτη που παρήγαγε φωσφορούχα λιπάσματα αλλά οδήγησε και σε εισαγωγή αζωτούχων λιπασμάτων από τη Ρωσία. Επίσης είχαμε 25 ε, δισεκατομμύρια ε, ευρώ τζίρο που και τελικά προτάθηκε 60 χιλιοστόγραμμα και ε, μια μεταβατική περίοδο πριν την επανεξέταση. Είναι υπερβολική η συμβαστική αυτή λύση, υπερβολικά φιλόδοξη και δεν στηρίζεται και από επιστημονικά πορίσματα να έχουμε τόσο δραστικές οριακέ τιμέ περιεκτικότητας καδμίδου. Άλλωστε, τα φωσφορούχα λοιπάσματα και τα ζωτούχα λοιπάσματα είναι πολύ ακριβά και ουσιαστικά υπονομεύουμε τη δική μα χημική βιομηχανία υπέρ των εισαγωγών από τρίτε χώρε. Εμεί είχαμε πολύ χαμηλότερα ποστά καδμίου, όπω φαίνεται ε, στην περιεκτικότητα του εδάφου μα σε καδμίο. Άρα δεν, ήταν επιζήμια η χρήση αυτών των λοιπασμάτων. Επίση, ε, και με τα οργανικά λοιπάσματα υπάρχει κίνδυνο ρήπανση ε, και λόγω τη χρήση αντιβιωτικών. και σίγουρα ε, μερικές φορές εισάγουμε προϊόντα από χώρες που έχουν πολύ χαλαρότερες προδιαγραφές και νομοθεσία. Δεν έχει αποδε... Ήταν πολύ δύσκολη η ολοποίηση αυτής της συμβαστική τροπολογία. γι' αυτό τελικά θα την υπερψηφίσουμε. Εκ μέρου των φιλελευθέρων. Κύριο κύριος Κατάινεν. Α, η κυρία Κατάινερ, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γεωργοί στο μέλλον ε, θα έχουν ε, ε, μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής προϊόντων. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον μας. Και το έδαφος, τα ύδατα, τα τρόφιμα δεν πρέπει να μολύνονται. Πρόκειται βέβαια και για την κυκλική οικονομία. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αν θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να προστατεύσουμε τη Βαλτική θάλασσα, ε, θα πρέπει να βελτιωθούν οι οριακές τιμές για το κάδμιο. Ε, το κάδμιο μπορεί να είναι επικίνδυνο για, τον, για την ανθρώπινη υγεία και γι' αυτό πρέπει να είμαστε αυστηροί. Εμείς στη Φινλανδία είμαστε πολύ αυστηροί σε σχέση με το κάδμιο για να προστατεύουμε καλύτερα τους ανθρώπους και τη φύση και ελπίζω αυτή την άποψη να τη συμμεριστούν και άλλες ε, και ε, και άλλα κρατημέλη. Κύριε Χόισλινγκ, ένα μισή λεπτό έχετε στη διάθεσή σα. Αγαπητοί συναδελφοί, ε, θέλω να σας πω ότι αυτή τη σημαστική πρόταση, ναι μεν τη δέχομαι, αλλά να σας πω και το εξή. Αυτή τη στιγμή έχουμε οριακή τιμή για το κάδμιο, τα 60 μιλιγκράμμ, αλλά πρέπει να σκεφτούμε από τι ξεκινήσαμε ως Κοινοβουλίο. Στην αρχή θέλαμε 40 με 20 στο Συμβούλιο, υπήρξε μπλοκάρισμα και λόγω οικονομικών συμφερόντων και τώρα καταλήξαμε σε μια πολύ ήπια συμβαστική λίστα έλεγα τα 60 μιλιγκράμμ. Αυτό λοιπόν θα, μας πρέπει, θα πρέπει να μας καταστήσει σαφές ότι την ώρα ε, που μπαίνουν τα λοιπάσματα στο έδαφος κάποια στιγμή θα αλλάξει και η διατροφική αλυσίδα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη συμβαστική πρόταση και χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αναγκασμένη μετά από κάποια χρόνια να αναθεωρήσει όλο αυτό το θέμα και να καταλήξει σε πιο φιλόδοξου στόχους. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα συμφωνήσουμε ε, γιατί εδώ και 30 χρόνια συζητάμε για το θέμα αυτό να που επιτέλους έχουμε έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα, κάτι και αυτό υπάρχει μια οριακή τιμή. Πρέπει όμω επίση να είναι σαφέ ότι αυτό το μπλοκάρισμα από πλευρά Συμβουλίου δεν ήταν καθόλου καλό. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο το Συμβούλιο φταίει που δεν προχωρήσαμε και δεν επιτύχαμε φιλόδοξου στόχου. Και να σα υπενθυμίσω και ότι η συνεργασία ανάμεσα στην ΙΜΚΟ και την ΕΝΒΗ δεν ήταν πάντα και η καλύτερη από αυτού του θέματο. Χρειαστήκαμε λοιπόν τρία ολόκληρα χρόνια για μια συζήτηση που τώρα πια, μπορούμε να την ολοκληρώσουμε, αλλά ξαναλέω και τονίζω, αυτή είναι απλά η αρχή. Γιατί στο τέλος πρέπει να καταλήξουμε στα 20 mg τιμή και όχι να παραμείνουμε στα 60. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος ε, Εκ έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Κυρία Πρόεδρε, η ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα από βιολογικές καλλιέργειες, η ζήτηση αυτή αυξάνεται συνεχώς. Και αυτό υπάρχει λόγος γιατί γίνεται έτσι. Οι άνθρωποι φοβούνται να δηλητηριαστούν από δηλητηριασμένα λιπάσματα. Το κάτμιο στα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες μέχρι και στο θάνατο. Αυτή λοιπόν η έκθεση σε κάτμιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλότερη από ό,τι μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ό,τι είναι πάνω από τα 20 μιλιγκράμμ ανά κιλό ε, κάτμιο, πάντα περιεκτικότητα κάτμιου. αυτό πρέπει να απορρίπτεται για λόγους υγείας. Η σύσταση της ΕΦΣΑ που λέει ότι ε, τα φωσφορούχα λιπάσματα είναι το βασικό έτμιο και για την επιβάρυνση με κάτμιο, αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Και όλες αυτές οι πληροφορίες οδήγησαν στο ότι ε, κάποιοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάλι ακολούθησαν τις ε, συστάσεις της ε, φαρμακοβιομηχανίας. Χάσαμε την ευκαιρία να αποφύγουμε την ρήπανση του περιβάλλοντος και του εδάφους. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με την πρόταση που κατατέθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τροστινσκή, από το Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, 50% των λοιπασμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά δεν έχουν ε, πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δώσουμε ένα τέρμα σε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό που προσβάλλει ένα ολόκληρο κλάδο που είναι πολύ ελπιδοφόρο για την γεωργία στην Ευρώπη. Οπότε για τα οργανικά λιπάσματα προσδιορίζει συνθήκε ίσου ανταγωνισμού με τα ανόργανα λοιπάσματα ορυκτή προέλευση. Και αυτό αποτελεί ένα αναπόσπαστο ε, τμήμα του πακέτου κυκλική οικονομία και καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλέ ε, παράπλευρε ανησυχίες και προβληματικέ γεωπολιτικού χαρακτήρα. Μερικοί δύσκολα συνδύασαν οικονομικά κριτήρια και κατάλληλη προθεσμία για συμμόρφωση στα νέα κριτήρια. Πάντως ε, τα αποτελέσματα της Διοργανικής Συμφωνίας κατέληξαν σε μια σωστή συμβαστική λύση που θα πρέπει να συμπληρωθεί για να τονώσουμε την καινοτομία στον τομέα παραγωγής λιπασμάτων και σκέφτομαι κυρίως ε, τη γαλλική χημική βιομηχανία που θα υποφεληθεί ιδιαίτερα από τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Τροστσίνσκι. Έχετε μία ερώτηση με μπλε κάρτα, κυρία Τροστσίνσκι, από τον κύριο Άγνιου. Τη δέχεστε? Yes. Would my colleague agree that where... Συμφωνεί ο συνάδελφος ότι ενώ το κάδμιο ε, είναι ε, στα φωσφορικά ε, είναι ασφαλές. Αν όμως εξορίσετε, τότε η συγκέντρωσή του αυξάνεται, γίνεται τοξικό και δεν μπορεί να ε, απομακρυνθεί εύκολα. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Δίκιο έχετε. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει κάπου, όλα γίνονται τοξικά ως διαμαγείας. Στη συγκεκριμένη μου περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όντως οι συνέπειες της νέας νομοθεσίας ε, δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμη. Ελπίζουμε πάντως ότι στη συνέχεια θα διαθετηθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροζάτη το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός για τα είδη λίπανσης ε, ανοίγει την αγορά σε νέα προϊόντα, κυρίως οργανικά λιπάσματα και ανόργανα λιπάσματα ορυκτής προέλευσης. Με ικανοποίηση διατυπώνω ότι απομακρυνθήκαμε από τις υπερβολικά δραστικές, ε, πολύ χαμηλές και δικαιολόγες ορικές τιμές ε, περιεκτικότητας καδμίου στα φωσφορούχα λιπάσματα. Θέλουμε να, τονίσουμε, να τονώσουμε το κλάδο μας και να εξασφαλίσουμε γεωργία με ασφαλή προϊόντα. Τελικά τα 60 χιλιοστόγραμμα ε, που είναι η συμβαστική λύση για το κάδμιο, συγχαίρω τον εισηγητή του οργάνου, εξακολουθούν να είναι υψηλέ ε, ε, οριακέ τιμέ που επηρεάζουν το κόστο τη παραγωγή. Και αυτό δεν αφορά μόνο την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, αλλά και άλλε τεχνικέ προδιαγραφέ που επιβάλλονται στην παραγωγή λιπασμάτων. Ε, θα έχουμε υπερβολικά, υπερβολικές συνέπειες για τον τομέα αυτό, αλλά και για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Επίση, σε ό,τι αφορά τα οργανικά λοιπάσματα που μερικέ φορέ χρησιμοποιούνται από δευτερογενείς πρωτεσίλες, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση μη κατάλληλων γεωπονικών προϊόντων μόνο χάρη αύξηση της αποδοτικότητας ε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τελικά το κόστος παραγωγής έχουμε προβλήματα με τα λοιπάσματα που θα επηρεάσουν και τους καταναλωτές. Γι' αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε ε, την αγορά λοιπασμάτων με γνώμονα την ε, υγεία του καταναλωτή, αλλά και την ανάγκη ασφάλισης ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων καθ' όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιλέρα Γκαρσία από τους Σοσιαλιστές. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω στη συζήτηση με κάποιες παρατηρήσεις. Μιλούμε για έναν κανονισμό που εντάσσεται στο πακέτο κανονισμών για την κυκλική οικονομία και που θα τεθεί σε ισχύ 20 χρόνια μετά τον ισχύοντα κανονισμό με σημαντικές αλλαγές και απαραίτητες επικαιροποίησεις. Τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη γεωργία. Μπορεί όμως να έχουν σημαντικούς κινδύνους ή αρνητικό επιζήμιο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Και αυτές τις αρνητικές συνέπειες θέλουμε να διορθώσουμε τον νέο κανονισμό. Πολλοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμπερίληψη και των οργανικών λοιπασμάτων. Όντως, αλλά για τα οργανικά λοιπάσματα, είναι να πούμε κάτι. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την καινοτομία, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους και σίγουρα να γίνουν σεβαστές ε, οι απαιτήσει της οδηγίας ε, για την ητρορύπανση και για τα οργανικά λοιπάσματα. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω, εγώ είμαι υπέρ της συμβαστικής λύσης για το κάδμιο. Η συμβαστική λύση ήταν ισορροπημένη και σε αυτά τα 60 μιλιγκράμμ, τα 60 χιλιοστόγραμμα, καταλήξαμε σε μία συμφωνία συμβιβαστική όπου όλοι έκαναν υποχωρήσεις. Και αυτή η μείωση νομίζω ότι είναι κατάλληλη, αυτή η ωριακή τιμή είναι κατάλληλη και ανταποκρίνεται στις παρούσες μας ανάγκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Ντεκάστρο τώρα. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα λοιπάσματα ποιότητας ε, ήταν και θα είναι πάντα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη πιο παραγωγικών μοντέλων παραγωγής. Ε, στο μέλλον θα πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ε, για τα τρόφιμα. Πρέπει να παράγουμε περισσότερο, όμως με μικρότερη ρήπανση. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Ταραμπέλα για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε και τον εισηγητή βέβαια για τη δουλειά τους για θέματα εναρμόνιση και θέματα σήμανση των λοιπασμάτων. Καθόρισαν πολύ φιλόδοξου στόχου όσον αφορά τη ρήπανση και κινητροδότησαν την έρευνα προ όφελο των γεωργών μα, όλα αυτά αλλά κυρίω όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Οι διαπραγματεύσεις δείχνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προηγείται στη βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργούν οι απαραίτητες προποθέσει, έτσι ώστε να έχουμε όλο και πιο καινοτόμα προϊόντα, αποτελεσματικά προϊόντα, που δεν θα επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον, θα εντάσσονται πολύ καλά μέσα στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Πολύ ωραία. Ε, τώρα λοιπόν θα ξεκινήσει η διαδικασία Catch the Eye. Ε, δύο ομιλητές, ε, σε δύο ομιλητές θα δώσω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι χάσαμε μια ευκαιρία για την κυκλική οικονομία στη Γεωργία. Εργάζομαι πάνω σε αυτό το θέμα, ε, ανόργανα λοιπάσματα από ε, και ε, από κοπριά. Ε, θα πρέπει να υπάρχει κατεξουσιοδότηση πράξη για την αναγνώριση ε, των προϊόντων αυτών των λιπασμάτων ως πράσινα λιπάσματα. Είχαμε μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιμένουμε μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θυμίζω και την απόφαση των Υπουργών που ε, είπαν ότι θα ε, δεχθούν τα λοιπάσματα αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Σιόιντροβα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον ε, ε, εισηγητή, τον για τη συμβιβαστική λύση που καλύπτει τους γεωργούς και όσους ενδιαφέρονται για ασφαλή τρόφιμα και ασφαλές περιβάλλον. Χαίρομαι για τα κατώτερα επίπεδα ε, του καδμίου. Αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια του περιβάλλοντος και του εδάφους βέβαια. Μιλήσαμε πολύ για τη μόλυνση των υπογείων υδάτων από τις χημικές ουσίες, τα λοιπάσματα. Η νομοθεσία αυτή θα βοηθήσει προς ε, την επίλυση αυτού του προβλήματος. Δεν θα είναι πια αναγκαίο να ε, ε, καταγράφονται ε, ε, τα προϊόντα σε, με βάση διαφορετικούς κανονισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο λεπτά ο κύριος Τίμερμανς. Κυρία Πρόεδρε, ε, μία συγκεκριμένη ερώτηση που θέλω να την απαντήσω. Η, η έκθεση για τη μελέτη θα είναι έτοιμη πριν από το τέλος του έτους. Οπότε δεν θα περάσει πολύς χρόνο μέχρι ότου ενημερωθείτε. Και επειδή είναι ευρύτατη η μελέτη, έχουμε αρκετέ εγγυήσει για να υποθέσουμε ότι θα πάει προς την σωστή κατεύθυνση που θέλετε κι εσείς. Παρακολουθείτε το θέμα και όταν είναι έτοιμη η μελέτη θα τη δείτε. Ε, κατά τα άλλα θα ήθελα να πω ότι η εξέλιξη αυτή είναι καλή για τους γεωργούς, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το περιβάλλον και πάνω απ' όλα είναι καλός ο κανονισμός για την υγεία μας. Κάναμε ακόμα ένα βήμα μπροστά, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα για μελλοντικά βήματα στο μέλλον. Ε, το, το, η εργασία μας ε, σήμερα μας οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρέοδρε για την προσπάθειά σας και για, τη... για το σημαντικό έργο που έκανε η ομάδα σας. Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα, το λόγο έχει για δύο λεπτά ο εισηγητής ο κύριος Τουρκάνου και συγχαρητήρια και πάλι για την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Τίμερμανς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλια που έκαναν και να πω στους κυρίους Ταραμπέλα Τσέσχακ, Ιβάσκοβιτς, Κάλλας, Δάρεν Μαστάλκα, Χαϊτεμα και φυσικά και στην κυρία Καρτίνη. Θερμά ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για το θέμα των ειδών λίπανσης. Όπως είπε κάποιος συνάδελφος, διαπιστώσαμε ότι ήταν ε, καλές και ισορροπημένες οι διοργανικές διαπραγματεύσεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας ε, ζητήσω να υπερψηφίσετε ομόφωνα την έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τουρπάνο. Σας συγχαίρω και εγώ για την προσπάθειά σας και την ε, έκθεσή σας. Ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό και θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. al Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μια έσταση εδώ, βάσει του άρθρου 182 του Συντερικού Κανονισμού. Θα ήθελα να θέσω ένα διαδικαστικό για την εγκυρότητα της ψήφου το, στο 108-2018 την ψηφοφορία στην, της έκθεσης νομικής επιτροπής για την πνευματική διοκτησία στην ενιαία αγορά. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της έκθεσης αυτής της Γιούρη, 312 ε, ε, ψήφισαν υπέρ σε μία ψηφοφορία και μετά τον το ελέγξαμε ότι, και είδαμε ότι 13 ευρωβουλευτέ άλλαξαν γνώμη και θέλουν να ψηφίσουν υπέρ σε μια ξεχωριστή ψηφοφορία μια τροπολογία. Θα ήθελα επίση να ζητήσω από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να επαναλάβει αύριο την σχετική ψηφοφορία. Γιατί ήταν σαφέ ότι κάποιοι ευρωβουλευτέ άλλαξαν γνώμη και αποφάσισαν να ψηφίσουν διαφορετικά. Υπήρξε μια παραπλάνηση του στη διάρκεια τη ψηφοφορία και θα ήθελα να αλλάξει το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Θέλω όμως να σας ανακοινώσω ότι με βάση τον εσωτερικό οργανισμό οι διορθώσεις ψηφοφορίας δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δηλαδή ό,τι ακολουθεί μετά την ψηφοφορία αυτό μπορεί να γίνει ε, το ξέρετε αυτό. Και κατόπιν αυτές οι αλλαγές ε, καταγράφονται, δημοσιεύονται, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αυτά λέει ο κανονισμός μας. Ε, κατόπιν τούτου το αίτημά σας θα το στείλω στο Προεδρείο, αλλά φοβάμαι ότι ο κανονισμός επ' αυτού του θέματος είναι απόλυτα σαφής. Αν δεν υπάρχουν άλλα διαδικαστικά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε πάρα αυτά με τις ψηφοφορίες. Πρόκειται Ξεκινάμε. Ε, έκθεση Winter Swibon, πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίαση κεντρικών αντισυμβαλόμενων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Σουίμπορν. Παρακαλώ, κυρία Σουίμπορν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, οι υποφαινόμενοι και η εισηγητρία επαναφέραμε το θέμα αυτό για την τελική ψηφοφορία γιατί οι διοργανικές διαπραγματεύσεις που είχαμε ε, ελπίσει να ξεκινήσουμε πριν από ένα χρόνο δεν έχουν ξεκινήσει ούτε τώρα. Ε, θέλουμε προτεραιότητα σε αυτό το σημαντικό θέμα που είναι απαραίτητο για την ε, μελλοντική χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη ενιαία αγορά. Ο κανονισμό αυτό στόχο έχει να αποτρέψει ε, τον κίνδυνο συγκέντρωση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγει κάποια ακραία σενάρια, εξασφαλίζοντα την ανάκαμψη και την